πολύ, κυρία Μογκερίνη. Τώρα λοιπόν έχετε και το λόγο για να κάνετε την ε, καταληκτική σας παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατανοώ ότι είμαι η μόνη στις ακροάσεις που δεν σας έδωσε ούτε σε εσά ούτε ε, στους διερμηνείς κάποιο γραπτό κείμενο. Ε, για την αναρκτήρια ομιλία μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχω σχεδόν τίποτα και για την ε, κατακλίδα της παρέμβασής μου. Θα είμαι πολύ σύντομη. Απλά θέλω να πω ότι σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για τις τρεις ώρες και κάτι που μου αφιερώσατε που ήταν ιδιαίτερα πολύτιμος αυτός ο χρόνος για μένα ε, για να μπορέσω να προετοιμαστώ για τη δουλειά μου, αν βέβαια συμφωνείτε κι εσείς, και για να μπορέσω να κατανοήσω καλύτερα τις απόψεις σας και τις ε, προτεραιότητές σας. Νομίζω ότι μπορούμε να δουλέψουμε θαυμάσια στο μέλλον και ομολογώ εξεπλάγει ότι για το ότι δεν ετέθησαν ερωτήσεις για τις ε, σχέσεις ε, που θα έχω με το Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω ότι πάρα πολλά ήδη ε, τα έχω γράψει στο ερωτηματολόγιο μου, αλλά θέλω να σας πω ότι θα μου άρεσε πάρα πολύ να έρχομαι όσο πιο συχνά γίνεται στο Κοινοβούλιο και νομίζω έχει γίνει πρόταση να συναντιόμαστε πριν και μετά από συγκεκριμένες συναντήσεις πριν από συναντήσεις ε, του ε, Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Προφανώς ε, λοιπόν οι ερωτήσεις είναι όλες νόμιμες, αλλά για μένα τουλάχιστον θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να συναντιόμαστε πριν από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Και επίσης θα ήθελα να γίνεται και μία εκ των υστέρων συζήτηση για τις συναντήσεις της Ειδικής Επιτροπής. Ξέρω ότι και εσείς μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να δουλέψουμε ένα ρεαλιστικό τρόπο και θα ήθελα επίσης ε, να πω και κάτι που ε, δεν αναφέρθηκε σχετικά με το σύστημα εκχώρησης αρμοδιοτήτων. Ε, με τον κύριο Γιούνκερ και με τους επιτρόπους ε, εγώ θεωρώ ότι όταν υπάρχει ένα θέμα σημαντικό μπορώ να ζητήσω από τον Επίτροπο κύριο Χάν να αναλάβει κάποιο θέμα. Ε, νομίζω ότι πρέπει να διαρθρώσουμε κάπως τη δουλειά μας, τη συνεργασία μας και όπως σας είπα θα είμαι ιδιαίτερα ευτυχή στο να ε, αναλάβω πρωτοβουλή στον τομέα της κοινοβουλευτική ε, διπλωματία. Το έχω κάνει αυτό και ε, είναι κάτι που το εκτιμώ ιδιαίτερα. Πάνω σε αυτό λοιπόν θα ήθελα επίσης εάν τελικά αναλάβω το αξίωμα της ΥΠΑ της εκπροσώπου, θα ήθελα όλα αυτά να τα μοιραζόμαστε για να είναι όσο πιο επωφελή γίνεται. Και θεωρώ ότι ιδιαίτερα σημαντική είναι και η ανταλλαγή απόψεων με τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών, με τους ειδικούς απεσταλμένους. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να το ενθαρρύνω αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να βρούμε κάποιους τρόπους ε, έτσι ώστε η Επιτροπή να μπορεί να έχει πρόσβαση ε, σε πολιτικές εκθέσεις, να βρούμε κάποια διαρθρωμένη μορφή συνεργασίας. Είπα στην αρχή, πιστεύω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να είναι το κέντρο αναφοράς όλων των εξωτερικών δράσεων ε, των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμών. Προφανώς και εννοούσα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τελειώνοντας λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Και η σημερινή συζήτηση κατέδειξε ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Αύγουστο, το πρώτο που είπα ήταν ότι γνωρίζω οι προκλήσεις είναι τεράστιες και κάθε μέρα ε, συνειδητοποιώ ότι είναι ακόμα πιο τεράστιες οι προκλήσεις από ό,τι πίστευα. Πάντως θεωρώ ότι έχουμε πέντε χρόνια μπροστά μας για να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις προκλήσεις. Ε, οι φιλοδοξίες είναι υψηπετής, μπορούμε να τις χαμηλώσουμε λιγάκι αν θέλετε, αλλά μέσα από την ε, συναδελφική ομαδική εργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και με καλές ε, μεθόδους ε, εργασίας, με ισχυρή πολιτική βούληση και ελπίζω και κάποιο καθοδηγητικό πνεύμα, ε, θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις στα θέματα που θίξαμε σήμερα εδώ. Μας περιπτώσει, εγώ υπολογίζω, προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας και στην υποστήριξή σας. Και όπως σας είπα, δεν είναι θέμα καθήκοντος αυτό, είναι θέμα πολιτικού συμφέροντος. Γνωρίζω ότι στο Κοινοβούλιο πολλά από αυτά που είπα εγώ τα εσημερίζονται και πάρα πολλοί άλλοι. Κυρία Μογκερίνη, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν αρκετά ακριβής έτσι και ευσύνοπτη η συνεδρίαση. Ε, εγώ ε, σας ευχαριστώ πολύ και για τις γραπτές σας απαντήσεις και αυτό το τελευταίο που είπατε για ποιο τρόπο θα βρούμε για να διαρθρώσουμε τη συνεργασία μας και να τη βελτιώσουμε κοινοβουλίο με τις δικές υπηρεσίες και μεταξύ αυτών εκτός από τις δυνατότητες ελέγχου και εκ των προτέρων διαβουλεύσεων για στρατηγικές συμφωνίες και σε άλλες σημαντικές αποφάσεις έχει σημασία ανταλλαγή πληροφοριών. Το θέμα αυτό με τα διαφημισμένα έγγραφα και πολλά άλλα ακόμα τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές πιστεύω ότι και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δομή και διάρθρωση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης ε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ακούστηκε, και οι συμφωνίες που έχουν γίνει, πούμε η συμφωνία της Μαδρίτης, σε κάποιους τομείς ε, εξακολουθούν να έχουν προβλήματα και χωλαίνει η εφαρμογή τους. Για να δούμε λοιπόν με ποιο τρόπο θα ανταποκριθείτε σε αυτά τα ζητήματα. Και μεταξύ αυτών ε, είναι και κάποια που έχουν να κάνουν με τη λύση του 1 τρίτο, 1 τρίτο, 1 τρίτο ή το θέμα της μείωσης των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων που έχουν και σχέση με τους ειδικού απεσταλμένους. Τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν ή τις συνολικές αντιμετωπίσεις, ε, τη λύση των κρίσεων. Αναφερθήκατε κι εσείς μπορούμε να τα συζητήσουμε περισσότερο. Και ακριβώς να έχουμε αυτή τη συνέργεια και το αποτέλεσμα μεταξύ των τριών Ευρωπαϊκή Δράση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. και να αναπτύξουμε όπως οφείλουμε ένα περισσότερο ομαδικό πνεύμα μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Και εσείς δηλώσατε προθυμία να ε, παίξετε ένα ρόλο ενεργού ε, αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ που απαντήσατε και δεσμευτήκατε σε όλα αυτά τα θέματα. Τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε και με τα δημοσιονομικά και πώς θα τα ξεκαθαρίσουμε. Και με τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού ενδεχομένω έχουν να κάνουν αυτά και θα πρέπει και ε, στα οικονομικά μας να είμαστε αποτελεσματικοί γιατί λόγω κάποιων κανόνων που οι ίδιοι επιβάλαμε σε αυτούς μας είναι ένας γραφειοκρατικός κορσές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και υποβληθήκατε σε αυτό το ε, ε, εγχείρημα της ακρόασης των ερωτήσεων. Απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις και ελπίζω να αναπτυχθεί έτσι μια συνεργασία και ελπίζω και γενικά αυτό να ισχύει για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αύριο το πρωί στις 8, στις 9 μάλλον, 9 αύριο το πρωί στο διευρυμένο Προεδρείο θα ασχοληθούμε με την επιστολή που θα πρέπει να γράψουμε για την αξιολόγηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Καλό σας βράδυ.